Συμβουλίου κινητήρια δύναμη για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών τους, ώστε να μπορούν να ζουν σε μια Ευρώπη που πραγματικά φροντίζει για την ασφάλειά τους. Σα ευχαριστούμε θερμά. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε τώρα. Η ψήφιση θα γίνει αύριο το μεσημέρι, 12 το μεσημέρι. Η ψήφιση της έκθεσης. Αξιότιμοι συνάδελφοι, επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι και ακολουθεί τώρα η κοινή συζήτηση για τη συμφωνία επανεισδοχής. Αφενός για τη σύσταση του κυρίου Τσάμπα Σόμπορ για την επανεισδοχή όσον αφορά ΕΕ Πακιστάν και δεύτερον για την ερώτηση, προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ε, αναμένουμε να απαντηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συμφωνία επανεισδοχής με τρίτες χώρες. Πρώτος που θα παρέμβει είναι ο κύριος Σόγκορ ως εισηγητής. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ. érvénybe Μιλάμε για την πρώτη συμφωνία επανεισδοχής με την οποία καλούμεθα να συμφωνήσουμε. Το Συμβούλιο έδωσε συγκεκριμένη εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακιστάν. Η εντολή αυτή δόθηκε στα τέλη του 2000 και τελικά υπεγράφει η συμφωνία αυτή τον προηγούμενο Οκτώβριο του 2009 μετά από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον διάδοχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που προϋπήρχε και γι' αυτό θα πρέπει να συμφωνήσει εκ νέου. Η γνώμη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων είναι θετική, εξίσου θετική είναι επίσης και η Επιτροπή οι υπόλοιπε επίσης αρμόδιες επί της ουσίας επιτροπές. Στόχος της Συμφωνίας Επανεισδοχής είναι να επιταχυνθούν οι συμφωνίες αυτές ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Δημοκρατία του Πακιστάν. Υπάρχει υποχρέωση πλέον για τη διαδικασία αποδοχής της ε, επανεισδαχής της νομικής αυτής ρύθμισης. Είναι ένα σημαντικό μέσο νομίζω για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και της διασφάλισης ε, των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πακιστάν είναι χώρα και διαμετακόμισης και προέλευσης μεταναστών οι οποίοι πολλές φορές έρχονται ε, χωρίς να έχουν το δικαίωμα αυτό για να ζήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία με το Πακιστάν λοιπόν είναι μια συμφωνία η οποία έχει και περιφερειακό βάρος θα έλεγα διότι θα διευκολύνει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να έχει στενότερες σχέσεις με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στη συμφωνία αυτή επανεισδοχής θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη διεθνή τάξη, νομική τάξη και το Πακιστάν καλείται πλέον να σεβαστεί τους, διεθνούς, τους διεθνείς συγγνώμη, κανόνες. Δημιουργείται μια συγκεκριμένη επιτροπή. Ε, στην επιτροπή αυτή, την μεικτή επιτροπή επανεισδοχής, συμμετέχει μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνει το Κοινοβούλιο τακτικά για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Επανεισδοχής. Και έχουν πλέον ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επικύρωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προσπάθεια που έκανε, όπως επίσης και τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους και ελπίζω να ψηφίσουν υπέρ της συγκεκριμένης πρότασης. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα οι συντάκτες της ερώτησης. Ο κύριος Μωράης πρώτος, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Ζόμπορ για την προσπάθεια που έκανε. Είχαμε καταψηφίσει την πρόταση αυτή στην αρχή για δύο λόγους. Πρώτον και για τα θέματα ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύουμε ότι στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής δεν, ε, γίνεται, δεν υπάρχει απόλυτος σεβασμός είτε τη σύμβαση της Γενέβης του 1951 και γενικότερα των δικαιωμάτων των μετανοστών. Όταν ε, υπογράφουμε τέτοιου είδους συμφωνίες θα πρέπει οι συμφωνίες αυτές να καλύπτονται από το διεθνές δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει ε, σε πολλές τέτοιου είδους συζητήσεις. Με τη Γεωργία και το Πακιστάν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και με την Τουρκία θα ε, υπογραφεί πάρα πολύ ε, σύντομα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει πάρει μέρος στη διαδικασία αυτή σε καμία περίπτωση. Οι απόψει του Κοινοβουλίου όμω θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν διαπραγματεύεται τέτοιου είδου συμφωνίε. Δεν πρέπει να αναμένετε ότι θα θα εμεί τυπικά και μόνο να επικυρώσουμε τη διαδικασία στο τέλο τη, όταν έχει ολοκληρωθεί. παρά την ε, πρώτη τέτοια συμφωνία η οποία τέθηκε σε ισχύ του 2004 δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ε, των ε, συμφωνιών αυτών. Και γι' αυτό ακριβώς η Σοσιαλιστική και Δημοκρατική Ομάδα ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε μια αξιολόγηση του μέτρου αυτού. Θα πρέπει να υπάρξει η διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων Θυμίζω ότι δεν έχει υπογράψει το Πακιστάν την σύμβαση της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Είναι μία από τις λίγες χώρες που δεν έχει κάνει και αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια κυρία Φλότρα, δύο λεπτά και εκείνη παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι ο εισηγητής μας δεν υπήρξε ειδικά αρκετά προσεκτικό ζητώντα μα να εγκρίνουμε μια συμφωνία που είναι ιδιαίτερα προβληματική. Πρώτον, μιλάμε για το Πακιστάν, όχι οποιαδήποτε χώρα. Το Πακιστάν είναι η χώρα η οποία επιδέχεται τον υψηλότερο αριθμό προσφύγων ήδη και θα του ζητήσουμε τι. Θα του ζητήσουμε να επιτρέψει την επανεισδοχή Πακιστανών αλλά Αφγανών και άλλων που είναι εδώ στην Ευρώπη και προσπαθούν να αποφύγουν ένα πόλεμο που εμείς έχουμε ξεκινήσει στο Αφγανιστάν. Πράγματι, το Πακιστάν δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση της Γενέβης και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Συμβουλίου της Ευρώπης μας ζητάμε να επικυρώνουμε συμφωνίες επανεισδοχής μόνο με χώρες που θα μπορούν να εγγυηθούν ορισμένα σημαντικά δικαιώματα σε θέματα προστασίας και υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά θέματα. Αν έπρεπε αύριο να ψηφίσω δεν θα ξέρα τι να κάνω. Ορισμένα άρθρα μπορεί να ε, αφορούν από 20 μέχρι 20.000. Γιατί? Γιατί κανένας δεν μας λέει τι απάντηση θα δοθεί σε αυτό στις αρμόδιες επιτροπές επανεισδοχής το άτομο ποιος θα μπορέσει να πει αν κάποιος να αποδείξει αν κάποιος έφτασε μετά την υπογραφή της συμφωνίας επανεισδοχής θα συμβεί μετά από την προθεσμή των 30 ημερών εάν δεν αντιδράσει το Πακιστάν και δεν χορηγήσει ταξιδιωτικά έγγραφα Μπορούμε λοιπόν να δεχθούμε αυτό το περίεργο κείμενο της, ε, της, της Ευρωπαϊκής άδεια Διέλευσης. Ξέρω ότι ούτε και εσείς δεν μπορέσετε να μου δώσετε απάντηση, κυρία Επίτροπε. Ούτε ο πρέσβης, ούτε ο πρέσβης του Πακιστάν. Δεν μπορώ λοιπόν να πω ότι συμφωνώ με αυτή τη συμφωνία εφόσον δεν είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας. Όλα θα εξαρτηθούν από τις απαντήσεις που θα δοθούν στα ερωτήματα αυτά. Γι' αυτό αύριο πρέπει να πούμε όχι σε ευχαριστώ. Κύριο κύριος δύο λεπτά και αυτός, επόμενος αγορητή. Ε, για αυτή την συμφωνία επανεισδοχής με το Πακιστάν. Νομίζω υπάρχουν προβλήματα ανάλυσης που πρέπει εδώ να ληφθούν υπόψη. Εδώ σε ένα επίπεδο μπορεί να δημιουργηθεί ένα επίπεδο μιας πρώτης συμφωνίας ε, για αυτού του είδους συμφωνίες ε, μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Εδώ υπάρχει ένα θέμα κοινοβουλευτικού ελέγχου και εξέτασης κοινοβουλευτικής που πρέπει να ληφθεί σε πολύ μεγαλύτερο βάθος υπόψη από ό,τι μέχρι σήμερα. Εδώ λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους αμφιβολίες και να υπάρξει αποσαφήνιση αυτών των θεμάτων για επόμενες συμφωνίες ε, όταν θα έρθει η ώρα να εγκριθούν από αυτή την Ευρωβουλή. Να υπάρχει πολύ πιο ενισχυμένη η διάσταση του ελέγχου και της εξέτασης στο κοινοβουλευτικό επίπεδο σε σχέση με τις ε, αρχές που ασχολούνται με τους ε, μετανάστες. Από την άλλη πλευρά αυτή η συμφωνία με το Πακιστάν δημιουργεί πολλές αμφιβολίες ε, σε σχέση με μια συμφωνία που δεν είναι μόνο σε σχέση με την επανεισδοχή Πακιστανών αλλά είναι ένα θέμα επανεισδοχής γενικά. Εδώ τίθεται το θέμα μιας χώρας ε, που σε σχέση με την ε, Συμφωνία της Γενέβης ε, έχει διαφοροποιήσει τη θέση της. Εμείς ή θα υλοποιήσουμε και θα σεβαστούμε αυτή τη συμφωνία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ή δεν θα σεβαστούμε αυτή τη συμφωνία και θα υπάρχει ένα πρόβλημα. Εδώ πρέπει να δούμε και την περίπτωση των γυναικών και την άσκηση βίας βάρος των γυναικών. Και πρέπει να δούμε το τι πρέπει να γίνει από πλευρά των αρχών του Πακιστάν και πρέπει με αυτόν τον τρόπο να δράσουμε. Για να ολοκληρώσω θέλω να υπενθυμίσω απλά ένα πράγμα το οποίο πρέπει να αναφερθεί. Εδώ και λίγο καιρό συζητούσαμε το θέμα των πλημμυρών στο Πακιστάν που προκάλεσαν 21 εκατομμύρια εκτοπισμένων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους. Πιστεύω ότι υπάρχει εδώ από πλευρά ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ένα είδο, ε, πώ θα έλεγα, κινησμού σε σχέση με 15 μέρε μετά με την υπογραφή μια τέτοια συμφωνία σε σχέση με την επανεισδοχή ατόμων σε σχέση με το Πακιστάν. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια έχετε εσεί τον λόγο, παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, εξ ονόματος της ομάδας μου θα ήθελα να πω ότι βεβαίως είμαστε υπέρ για τις συμφωνίες επανεισδοχής σαν ένα σημαντικό μέσο για την καταπολέμηση της πλατρείας μετανάστευσης που φαίνεται σαν πιο αποτελεσματικό από έναν πολλαπλασιασμό διμερών συμφωνιών. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τρία πράγματα. Σε αυτό το νέο νομικό πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται συστηματικά και τακτικά για τι διαπραγματεύσει και για την υλοποίηση αυτών των συμφωνιών, εφόσον συναποφασίζουμε. Μέχρι σήμερα 11 συμφωνίε έχουν ήδη υπογραφεί, συναυθεί και ε, έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσει για 7 άλλε, χωρί να υπάρχει οποιαδήποτε αξιολόγηση αυτών των συμφωνιών. Και προτού υπογράψουμε νέε συμφωνίε, ήταν απαραίτητο να αξιολογήσουμε εκείνε που έχουν ήδη συναυθεί. Τέλο, ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τι εγγύησει μπορεί να δώσει η Επιτροπή σε περίπτωση που τρίτες χώρε δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση τη Γυναίκα, όπως θύμισαν ορισμένοι συνάδελφοι. Επαναλαμβάνω λοιπόν, ε, παρόλο που προσωπικά ε, είμαι υπέρ μια συμφωνία επανεισδοχής με το Πακιστάν, υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές ε, γκρίζες ζώνες που δεν έχουν εξαλειφθεί. Έστω και αν η Επίτροπος Μέλστρομ, την οποία ευχαριστώ για τη δήλωσή της, έχει δώσει εγγυήσεις από πλευράς σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της ε, συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις με το Πακιστάν, ότι θα υπογράψει τις σημαντικές συμβάσεις που δεν έχει ακόμα υπογράψει, έστω και παρόλο που μας έδωσε την εγγύηση ότι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα θα μπορούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης στην πράξη, γεγονός παραμένει ότι πρέπει να θέσουμε ως προϋπόθεση για αυτή τη συμφωνία την υπογραφή από το Πακιστάν της Σύμβασης της Γενέβης. Διότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι πρέπει να βρεθεί σωστή ισορροπία ανάμεσα στο στοιχείο της ασφάλειας για όλους μας και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όποιο και να είναι το σημείο του πλανήτη όπου βρίσκονται. Διότι αυτό, πάνω, σε αυτό, πάνω σε αυτά τις αρχές στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει τον λόγο. Κυρία Επίτροπε, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι το Πακιστάν είναι στην επικαιρότητα, ιδιαίτερα τον τελευταίο μήνα και όλοι λυπούμεθα για τις απώλειες ε, της ανθρώπινης ζωής που χαρακτηρίζουν την επικαιρότητα στη χώρα αυτή και κάναμε ό,τι μπορέσουμε, ό,τι μπορέσαμε μάλλον για να ελαφρύνουμε τη δυστυχία της χώρας αυτής και να τη βοηθήσουμε να ανοικοδομηθεί και να προλάβει περαιτέρω τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές. Συζητήθηκε το θέμα του Πακιστάν ήδη την τελευταία εβδομάδα στο Συμβούλιο. Να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών και τον εισηγητή για την εξαιρετική προσπάθεια και την υποστήριξη που έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από το μήνα Ιούλιο. Η συμφωνία αυτή επανεισδοχή εδώ και αρκετά χρόνια είναι ένα σημαντικό μέσο διαχείρισης των μεταναστικών μεταναστευτικών ροών. Η πολιτική της μετανάστευσης και του ασύλου, εφόσον θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι στους πολίτες, θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή ότι αυτοί που δεν έχουν ένα νόμιμο τίτλο να παραμείνουν σε μια συγκεκριμένη χώρα πρέπει να διευκολυνθούν να επιστρέψουν στη χώρα τους, ε, στην χώρα προέλευσης ε, ή στην χώρα διαμετακόμισης από την οποία έχουν έλθει. Και ορίζονται οι τρόποι με τον οποίο θα γίνεται αυτό. Με τον χρόνο συνδέονται φυσικά όλες αυτές οι συμφωνίες επανεισδοχής και είναι αναπόσπαστα στοιχεία της διαπραγμάτευσης που κάνουμε με τις χώρες αυτές για τα θέματα της μετανάστευσης. Θα συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις διαπραγματεύσεις αυτές σύμφωνα με την εντολή την οποία έχει λάβει μέχρι τώρα. Να αναφερθώ σε λίγες από τις ανησυχίες τις οποίες έθεσαν ορισμένοι συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τηρήσει πλήρως ε, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από το 280 τη Συνθήκης. Πλήρως θα ενημερώνει ε, ταχύτατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις της διαπραγματεύσεις και για τις καταλήξεις στις οποίες θα οδηγούμεθα στα πλαίσια των συμφωνιών επανεισδοχής. Και θα λάβουμε υπόψη πλήρως τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην διαδικασία ε, ε, αποδοχής των συγκεκριμένων αυτών προτάσεων θα δίνουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, σύμφωνα πάντα φυσικά και με τις αρχές της εμπιστευτικότητας, όταν τρέχουν οι διαπραγματεύσεις. Και όλα αυτά θα γίνονται στα πλαίσια των σχέσεων των κανονικών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι η πρώτη ενημέρωση, πλήρης, έχει γίνει in camera προς την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών στις 12 Ιουλίου και η κυρία Γκρίσπεκ αναφέρθηκε και στη δήλωση την οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε από κοινού πώς μπορούμε τη συνεργασία μεταξύ μας να την βελτιώσουμε. Όταν κάποιες χώρες δεν έχουν υπογράψει τη Συμφωνία της Γενέβης, ε, προφανώς και θα θέλαμε οι χώρες αυτές να το κάνουν, προσπαθούμε να πείσουμε το Πακιστάν να υπογράψει τη Σύμβαση της Γενέβης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμένει στις, ε, στην αξία που έχουν τα διεθνή μέσα για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διεθνή προστασία. Και είναι φυσικά στο κέντρο της πολιτικής μας. Για τον λόγο αυτό Έχουμε αναπτύξει και ένα ευρωπαϊκό δεδομένο για τη διεθνή προστασία στα πλαίσια της οδηγίας για τη χορήγηση ασύλου και ε, φυσικά και στην ε, πολιτική παλινόστησης ε, και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύονται από τη Σύμβαση της Γενέβης για τους μετανάστες και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι λοιπόν κανένας άνθρωπος, κανένας πολίτης ε, δεν θα πρέπει να μετακινηθεί από οποιαδήποτε χώρα εάν ε, είναι στόχος δίωξης, ε, καταστολής, έχει υποστεί βία ή κινδυνεύει να υποστεί βία στην χώρα στην οποία κανονικά θα πρέπει να επιστρέψει. Γι' αυτό λοιπόν κάθε χώρα θα πρέπει να ελέγχει τις αιτήσει χορήγησης ασύλου και ε, να επιτρέπει στο συγκεκριμένο ε, πρόσωπο να παραμένει στη χώρα αυτή νόμιμα έως ότου ληφθεί η τελική απόφαση για τη χορήγηση ημί του ασύλου. Η αρχή λοιπόν της ε, αυτή είναι κάτι το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα πλαίσια των συμφωνιών επανεισδοχής. Όλες οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν τη ρήτρα λοιπόν η οποία ζητά την προστασία όλων αυτών των επιπέδων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι συμφωνίες ε, αυτές ε, επίσης θα ήθελα να πω ότι υπονομεύουν αποτελεσματικά τις δραστηριότητες των δικτύων παράνομης μετανάστευσης. Ήδη η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για την παράνομη ε, μετανάστευση από το Πακιστάν υπολογίζει ότι ο κύκλος εργασίας αυτής της παράνομης δραστηριότητας μόνο από το Πακιστάν τα προηγούμενα χρόνια ανήλθε σε 1,5 δις εκατομμύρια δολάρια και γι' αυτό ζητούν τα Ηνωμένα Έθνη να υπάρξουν ε, συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων δικαστικών όπως επίσης και συμφωνίες επανεισδοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει υπόψη τα συμπεράσματα αυτά στις διαπραγματεύσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει αξιολογεί τα αποτελέσματα των υπαρχουσών συμφωνιών ε, ε, πανισδοχής και ε, αξιολογεί και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όλες οι χώρες με τις οποίες έχει υπογράψει η διευκολύνση στον τομέα της χορήγησης θεωρήσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ελέγχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θέματα αυτά όπου υπάρχουν αντίστοιχες τέτοιες συμφωνίες επανεισδοχής. Ε, υπάρχουν αντίστοιχες επιτροπές ελέγχου των διαδικασιών επανεισδοχής συλλέγουμε όλες τις πληροφορίες για την εφαρμογή των συμφωνιών αυτών όπου υπάρχουν. Δεν έχουμε ε, προς το παρόν σημειώσει σημαντικά προβλήματα και ούτε έχουν σημειώσει σημαντικά προβλήματα στα πλαίσια της λειτουργίας των συμφωνιών επανιστοχής ή ΜΚΟ. Παρότι το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για πάρα πολλές από αυτές τις χώρες. Κανένα σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές δεν θα πρέπει να αποστέλλεται πίσω αν αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο να υποστεί διώξεις, βασανιστήρια και απάνθρωπες ε, μορφές μεταχείρισης. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό δεν είναι διαδικασία της συμφωνίας επανεισδοχής, αλλά μιας παράνομης απόφασης την οποία έχει πάρει ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος. Όπως επίσης ζητήθηκε και στα πλαίσια του προγράμματος της Στοχόλμης στο Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος του χρόνου θα παρουσιάσει μια απλήρη αξιολόγηση του συνόλου των ισχυουσών συμφωνιών επανεισδοχής. Στα πλαίσια λοιπόν της συγκεκριμένης αυτής αξιολόγησης θα εξετάσουμε την πιθανότητα στην οποία αναφερθήκατε, να υπάρξει δηλαδή δυνατότητα βοήθειας προς αυτούς οι οποίοι ε, ε, έχει αποφασιστεί η διαδικασία, να εφαρμοστεί η διαδικασία αυτή στην χώρα επιστροφής. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι για να υποστηρίξουμε τη διαδικασία, θα τους αξιολογήσουμε, υπάρχουν οδηγίες οι οποίες είναι σε λειτουργία, σε ισχύ. Εμείς θα σας κρατήσουμε ενήμερους όσο μπορούμε καλύτερα και όπως αναφέρεται στη Γενική Συμφωνία την οποία έχετε μπροστά σας και στην ανακοίνωση η οποία έγινε δεκτή από την Επιτροπή ε, Δημοσίων Ελευθεριών τον μήνα Ιούλιο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά κυρία Επίτροπε. Για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ο κύριος Αλμπερτίνη, ένα λεπτό παρακαλώ. Grazie Presidente. Dopo μετά από 8 χρόνια από την αρχή των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πακιστάν καταλήξαμε επιτέλους σε μια συμφωνία για τη διαδικασία επανεισδοχής για αυτούς οι οποίοι ε, ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τα κατάλληλα χαρτιά. Ε, μας ζητήθηκε να διατυπώσουμε και μία γνωμοδότηση για τη συμφωνία αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην περιοχή γύρω από το Πακιστάν και στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα συζητήσαμε τα θέματα αυτά επί μακρόν. Υπήρξαν κάποιες ανησυχίες για την αστάθεια στην πολιτική κατάσταση και το πρόβλημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πακιστάν. Οι διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Πακιστάν δεν έχουν δώσει εγγυήσει για τον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων αυτών που έχουν ε, μπει στη διαδικασία επανεισδοχής προς το Πακιστάν. Δεν υπάρχει επίσης και μια πλήρης αξιολόγηση των 11 συμφωνιών που είναι ήδη σε λειτουργία. Απαιτείται λοιπόν ένα ξεκάθαρο πλαίσιο ε, για την διαδικασία επανεισδοχής με το Πακιστάν. Είναι κάτι το πάρα πολύ προτιμότερο θα έλεγα από τις μεμονωμένες ad hoc ενέργειες επανεισδοχής τις οποίες θα αποφασίζουν τα διάφορα κράτη-μέλη. Το άρθρο 16 θα δώσει εγγυήσει για τους ελέγχους αυτούς. Γι' αυτό επαναλάβω το αίτημα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για την επανεξέταση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξεπεράσατε κατά πολύ τον χρόνο σας. Ακολουθούν οι αγορητές εξ των κοινοβουλευτικών ομάδων. Για το ΕΛΚ, ο κύριος Μάνφρεντ Βέμπερ, 1,5 λεπτό παρακαλώ. Αξιότιμη Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν για το θέμα του Πακιστάν. Συζητούμε σε μια δύσκολη συγκυρία για το Πακιστάν αυτό το θέμα και υποστηρίζουμε την αλληλεγγύη υπέρ των ατόμων που επλήγησαν από τις θεομηνίες. Όπως ανέφερε ο κύριος Σόγκα πιο πριν, εγώ θα ήθελα καταρχήν για τα θέματα της ε, Συμφωνίας Επανεισδοχής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτα κράτη να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, είναι σκόπιμες και χρήσιμες και αναγκαίες αυτές οι συμφωνίες διότι στην Ευρώπη έχουμε ένα δίκαιο το οποίο ρυθμίζει τα θέματα μετανάστευσης. Όταν ρυθμίζονται τέτοια θέματα μετανάστευσης, οι παράνομοι μετανάστες πρέπει να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες. Το επόμενο λογικό βήμα είναι η απέλαση, επανεισδοχή. Έχουμε πολλές φορές ε, τους αριστερούς και τους σοσιαλιστές στο πλευρό μας ε, επιθεωρητικού επίπεδου. Όταν έρχεται η ώρα της πρακτικής εφαρμογής, πολλοί αρνούνται να κάνουν το τελικό βήμα και γι' αυτό έχουμε αυτή την κατάσταση. Δεύτερον, ε, θα πρέπει να τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εναλλακτική λύση σε τέτοιε συμφωνίε φυσικά δεν είναι το ότι εμεί έχουμε καλύτερε προδιαγραφέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά αν δεχθούμε να έχουμε 27 διαφορετικέ προδιαγραφέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τα κράτη-μέλη, τότε δεν θα μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Τρίτον, πώ μπορούμε την εταιρική σχέση με τρίτε χώρε να την διαμορφώσουμε σε ένα θελκτικό, ελκυστικό πλαίσιο. Ζητώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί όταν ε, θα έχουμε τον επόμενο γύρο ε, με τις τρίτες χώρε θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να συζητηθούν τα θέματα επανεισδοχής. Ή όταν έχουμε το θέμα της μετανάστευση σε νόμιμο πλαίσιο πρέπει τρίτες χώρε να είναι σε θέση να μας κάνουν κάποιες υπαναχωρήσεις για τα θέματα επανεισδοχής. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ, ολοκληρώσατε. Μετά για την Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ακολουθεί η κυρία Σιλβί Γκυγιόμ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, η καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στο Πακιστάν μας υποχρεώνει να βάλουμε για 15 μέρες την ε, συμφωνία επανεισδοχής με αυτή τη χώρα. Σήμερα η επιλογή μας είναι καθοριστική πώς θα εγκρίνουμε αυτή τη συμφωνία ενώ παραμένουν χωρίς απάντηση τόσα πολλά ερωτήματα και υπάρχουν τόσες πολλές απορίες. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για το θλιβερό ρεκόρ του Πακιστάν σε ό,τι αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά πρέπει να θυμίσουμε επίσης ότι δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση της ε, ε, Γενέβη για τους πρόσφυγες απάτριδες. Και το πρόβλημα είναι ότι η συμφωνία αυτή αφορά συγκεκριμένα τους Αφγανούς και το να ζητάμε από, την από το Πακιστάν να επικυρώσει τη σύμβαση της Γενέβης δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε κάτι ε, ξεκάθαρα ότι η υπογραφή της σύμβασης της Γενέβης και άλλων σχετικών πράξεων είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία. Υπάρχει και η αφιβολία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας με ένα πεδίο εφαρμογής και τεχνικές λεπτομέρειες που είναι πραγματικά ανεφελώδεις τόσο σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή επίση προσωπικών δεδομένων. Και πέρα από την εφαρμογή υπάρχει και η όλη διαδικασία ε, υπογραφής ε, αυτής της συμφωνίας και άλλων. Κατ' επανάληψη ζητήσαμε από την Επιτροπή να μα δώσει στοιχεία για τι συμφωνίε που έχουν υπογραφεί. Δεν έχουμε στοιχεία, τα στοιχεία που μα αναφέρετε σήμερα δεν επαρκούν. Πώ μπορούμε λοιπόν λογικά να δεχθούμε, να εγκρίνουμε τέτοια συμφωνία χωρίς να έχουμε μια αξιολόγηση των προηγουμένων ε, συμφωνιών όπω ζήτησε η Επιτροπή Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει τι υποχρεώσει του αν δεν ενημερώνεται στη διάρκεια από τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και εφαρμογή αυτών των συμφωνιών. Ως σύνομοθέτη, το Κοινοβούλιο έχει αναλάβει πολύ πιο σοβαρές αρμοδιότητες και ευθύνες ε, όταν μιλάμε για, εταιρείες, για συμφωνίες ε, ε, εταιρικής σχέσης με χώρες όπως η Λιβύη ή για συμφωνίες επανεισδοχής όπως με, χώρε χώρες όπως το Πακιστάν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί πρωτού αποφασίσουμε οτιδήποτε. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε για τον, τη συμμαχία των Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών η κυρία Βίξτρομ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, όπως πολλοί συνάδελφοι αντιλαμβάνομαι ότι η χρονική στιγμή της συζήτησης για τη συμφωνία επανεισδοχή με το Πακιστάν ίσως δεν είναι κατάλληλη μετά από τις τρομερές πλημμύρες του Αυγούστου. Όλοι είδαν τις φρικώδεις εικόνες των εκτοπισμένων και συμμεριζόμαστε τα δεινά του λαού του Πακιστάν. Αλλά μην πέσουμε στην παγίδα η συμφωνία επανεισδοχής είναι ένας τρόπος να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Πακιστάν και γι' αυτό τη συμφωνία αυτή πρέπει να την δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αφενός υποστηρίζουμε την νόμιμη μετανάστευση, από την άλλη θέλουμε να πατάξουμε την παράνομη μετανάστευση. Ευχαριστώ την Επιτροπή για τις εγγυήσεις που μας έδωσε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των συμφωνιών. Μας εξήγησε σαφώ ότι ασκείται πίεση στο Πακιστάν ώστε να υπογράψει τη Σύμβαση της Γενέβης και υπάρχει δέσμευση για ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις συνέπειες της εφαρμογής αυτών των συμφωνιών επανεισδοχής. Η ομάδα μας υποστηρίζει αυτή τη συμφωνία επανεισδοχής που συζητούμε σήμερα θέλουμε η Επιτροπή να απαντήσει θετικά ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις, τα αποτελέσματα αυτών των συμφωνιών. Γνωρίζω ότι το γεγονός ότι δεν έχει υπογράψει το Πακιστάν τη Σύμβαση της Γενέβης δημιουργεί πρόβλημα. Αλλά όλες, όλα τα κράτη-μέλη δεσμεύονται από τη Σύμβαση της ε, και από την Ευρωπαϊκή ε, Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Εάν διώξουμε άτομα των οποίων ε, ε, ε, ζητήσουμε την επιστροφή ατόμων των οποίων ή την επαναπρόθεση ατόμων των οποίων τα ανθρώπινα δικαιώματα κινδυνεύουν θα ήταν λάθος. Η μη επαναπρόθεση είναι κάτι που πρέπει να ισχύει πάντα και αυτές οι συμφωνίες είναι μια ανάγκη για να οργανώσουμε καλύτερα τη συνεργασία με το Πακιστάν. Για τους πράσινους παρακαλώ η κυρία Σαρζεντίνη 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια πολιτική. Στην πολιτική ασύλου, όσον αφορά την πολιτική ασύλου και σε σχέση και με την επανεισδοχή, θα πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να είναι σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει η Ευρώπη πολλούς ανθρώπους που δεν μπορεί να τους απελάσει απλά σε, στη χώρα προέλευσης. Έχουμε τη χώρα διαμετακόμισης ή και τη χώρα ε, ε, προέλευσης που πρέπει να διαφοροποιούμε. Τώρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα χωρίς να ανύπτουμε τις ε, χείρες μας ε, θεωρώντας ότι είμαστε αθώοι. Όταν έχουμε το θέμα της απέλασης ατόμων στην Ερυθρέα ή όταν έχουμε το θέμα Αφγανών ε, που απελάβνονται στο Πακιστάν, όταν προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο εμείς προσχηματικά να επιλύσουμε το πρόβλημα, λένε κάποιοι ότι θα έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα θελκτικότερο, ένα πιο ελκυστικό πλαίσιο για τις τρίτες χώρες. Δεν μου φαίνεται ότι αυτό είναι ιδιαίτερα ανθρωπιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών των ανθρώπων, ούτε είναι και η πιο σκόπιμη και πιο χρήσιμη πολιτική από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν απελάβνονται προ την Τουρκία αυτά τα άτομα, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια άτομα που μέσω τη Τουρκία προσπαθούν να καταλήξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, φτάσουν σε, ένα, σε μια χώρα όπου δεν επιτρέπεται να βρίσκονται εκεί. Και όλες αυτέ οι διαδικασίε είναι πάρα πολύ δαπανηρέ. Για την Ενωτική Αριστερά, ο κύριο Ντεζόν, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Γκούε είναι αντίθετη με αυτό το σχέδιο επανεισδοχής με το Πακιστάν. Δεν είναι το κατάλληλο μέσο και έρχεται μια, μια μη κατάλληλη στιγμή. έχουν καταστραφεί οδοί γέφυρες, η χώρα έχει γυρίσει δεκάδες χρόνια πίσω. Υπάρχουν πάρα πολλά εκτοπισμένα άτομα σαν αποτέλεσμα των πλημμυρών. Δεν έχουν χάσει τα πάντα οι άνθρωποι. Κάτω από τέτοιες συνθήκες λοιπόν περιμένουμε από την Ευρώπη να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Και τι βλέπουμε. Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή αποφασίζεται να υπογράψουμε μια συμφωνία πεντοκής με το Πακιστάν με αποτέλεσμα η Ευρώπη να στείλει ετούντες άσυλο ή παράνομους στο Πακιστάν. Αυτό νομίζω ότι δεν συμβαδίζει με, τις θεμελιώδεις, με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία πρεσβεύουμε. Το Πακιστάν δεν είναι μια σταθερή χώρα αυτό που ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο είναι το εξή. Τι σας κάνει να έχετε εμπιστοσύνη σε μια χώρα η οποία δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση της Γενέβης. Τι σας δημιουργεί εμπιστοσύνη και σας κάνει να πιστεύετε ότι το Πακιστάν θα προστατεύσει αυτούς τους πρόσφυγες. Οι εγγυήσει που προβλέπονται σε αυτή τη συμφωνία ανταποκρίνονται στις υποχρώσεις μιας χώρας έναντι μιας άλλης. Το μόνο που ακούσαμε ωστόσο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαπιστώσει κατά πόσο τηρούν τις υποχρεώσεις τους τα κράτη-μέλη δυνάμει της Σύμβασης της Γενέβης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά πώς θα τα επαληθεύσετε όλα αυτά. Θα στείλετε υπαλλήλου στο Πακιστάν όταν θα, τα, τα, θα τοποθετούνται, ε, θα επιβιβάζονται σε ένα αεροπλάνο, πόσο καιρό θα παρακολουθείτε την τύχη αυτών των ανθρώπων. Και αυτή η συμφωνία έρχεται μια πολύ ακατάλληλη στιγμή, γι' αυτό λέμε όχι σε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ για τους μη εγγεγραμμένους. Εσείς έχετε τον λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σε ένα πρόβλημα με την Τουρκία. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να υπογράψει μια συμφωνία επανειδοχής με την Τουρκία. Αλλά η χώρα αυτή παρεμποδίζει αυτή την προσπάθεια. Αυτή είναι μια παράδεκτη κατάσταση για δύο λόγους. Πρώτον, θα μπορούσαμε να αναμένουμε συνεργασία από μια χώρα που είναι, εμφανίζεται υποψήφια αντί να παρεμποδίζει το έργο μας. Η Τουρκία δεν είναι γείτονα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια χώρα η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο κοινοτικό σύνορο αλλά είναι μια χώρα διέλευσης και προέλευσης παράνομης μετανάστευσης και σας παραπέμπω σε ένα πρόσφατο υπόμνημα της, του Ευρωπόλ, της, του Eurojust και του Frontex που λέει ότι η Τουρκία είναι η κύρια χώρα διέλευσης για το εμπόριο της ηρωίνης προς τα Βαλκάνια με, από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν και μια ε, από τις βασικές πηγές ε, του οργανωμένου εγκλήματος από ό,τι αντιλαμβάνομαι σε ό,τι αφορά την Τουρκία είμαστε υποχρεωμένοι να διαπιστώσουμε ότι η τουρκική κυβέρνηση ε, καταλήγει σε όρους οι οποίοι είναι παντελώς απαράδεκτοι. Ενώ μιλάμε για διευκόλυνση διαδικασία των θεωρήσεων η Τουρκία αρχίζει να μιλάει για άνοιγμα συνόρων, για ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων, Τούρκων πολιτών κάτι που το, μόνο που θα κάνει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση αντί να τη βελτιώσει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ακολουθούν οι άλλοι εγγεγραμμένοι αγορητές. Ο κύριος Κουέλιο, 1,5 λεπτό πρώτος, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Μάρκστρομ, αγαπητοί συνάδελφοι. Συγχαίρω τον συνάδελφο Σόγκορ για την έκθεση που μας παρουσίασε. Η σημασία αυτής της έκθεσης ε, και σε σχέση με όλα τα θέματα αυτά καταδεικνύονται ότι χρειάστηκαν 10 χρόνια για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Αυτή η συμφωνία είναι σημαντική όχι μόνο για το Πακιστάν, αλλά επίση και για τη δική μα σχέση με τι άλλε χώρε τη περιοχή. Είναι θετικά αυτά τα στοιχεία για την καταπολέμηση τη παράνομη μετανάστευση. Η επιστροφή όμω οποιοδήποτε θα μπορεί να βασίζεται σε βάση με μια ατομική απόφαση σε σχέση με τι ευθύνε και υποχρεώσει που απορρέουν από διεθνεί συμβάσει. Το Πακιστάν χωρίς αμφιβολία είναι μια σημαντική χώρα προέλευσης ή διαμετακόμισης ατόμων σε κατάσταση που ε, δεν είναι ασφαλής. Και εδώ έχουμε και το θέμα των ε, συμφωνιών αλλά επίσης και το, ε, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστήριων καθώς επίσης και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δημιουργούνται πολύ σημαντικές αμφιβολίες για την ασφαλή επιστροφή πολλών ατόμων σε αυτή τη χώρα και θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη την προστασία θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρότι είναι επιθυμητά αυτά τα θέματα για τα κράτη-μέλη, δεν πρέπει να γίνονται όλα αυτά ad hoc. Μέσα σε ένα σαφέ πλαίσιο συνεργασία με το Πακιστάν πρέπει να γίνονται με την επιτήρηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση όλων αυτών των παραγόντων. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Φρασικόβα Μπενιόβα, 1,5 λεπτό. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συζητούμε εδώ το θέμα των συμφωνιών επανεισδοχής και πολλοί από εμάς ανησυχούμε για θεμελιώδη θέματα όσον αφορά την ασφάλεια των ατόμων που εμπλέκονται σε σχέση με την επανεισδοχή. Οι συμφωνίες επανεισδοχής δεν λαμβάνουν υπόψη αυτές τις πτυχές. Υποτίθεται ότι όταν συμφωνούν δύο χώρες και συνάπτουν μια συμφωνία θα πρέπει να είναι σεβαστές αυτές οι πτυχές. Όμως μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεισδοχής αυτά δεν είναι σεβαστά. Υπάρχουν ευρύτερες συμφωνίες, ένα ευρύτερο πλαίσιο που αφορούν θέματα συνεργασίας όπως και την ασφάλεια στον ανεφοδιασμό με ενεργειακά προϊόντα, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και έτσι οι συμφωνίες επανεισδοχής είναι ένα πολύ μικρό τμήμα του μοσαϊκού των σχέσεών μας με αυτές τις χώρες. Να μην αυτά Για προηγμένες χώρες οι συμφωνίες επανεισδοχής είναι ένας κομψός τρόπος να ξεφορτώνονται τους παράνομους μετανάστες τους οι προηγμένες χώρες εξαγοράζοντας, ας το πούμε έτσι, από πλευρά της χώρας ε, εισδοχής ε, που δέχεται αυτά τα άτομα με κάποια προτερήματα που τους παρέχονται, εμπορικά ή άλλα. Δεν υπάρχει κανένα ε, λόγος ούτε να υπάρχει η πολιτική βούληση ούτε η ικανότητα από πλευρά της χώρας επανεισδοχής να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των ε, απελαυνομένων με αυτόν τον τρόπο. Για μας που ανησυχούμε για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει υπό το πλαίσιο των συμφωνιών επανεισδοχής και γι' αυτό τα θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων πρέπει να συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ. Νίλσεν. Κάθε απόφαση απέλαση που λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές μια συγκεκριμένη χώρας θα πρέπει να σέβεται το πρωτόκολλο του 67 τη σύμφαση τη Γενέβης και της διεθνή Συνθήκης. Κανένας δεν μπορεί να απομακρυνθεί προς μια άλλη χώρα όταν υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι, όταν κινδυνεύει να, όταν υπάρχει ε, θανατική ποινή και ε, απάνθρωπη μεταχείριση. Στο Πακιστάν υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θανατικές εκτελέσεις, εγκλήματα τιμής, ε, πολλές διεθνείς συμβάσεις δεν έχουν υπογραφεί. Πώς μπορούμε λοιπόν να ξέρουμε ότι τα άτομα που θα περάσουν από τη διαδικασία αυτή θα τύχουν σεβασμού των δικαιωμάτων της. Δεν υπάρχουν καθόλου εγγυήσεις για τις θρησκευτικέ και αφιλετικές μειονότητες, για τις γυναίκες, για τους Αυγανούς πρόσφυγες. Δεν υπάρχει ε, παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας αυτής από πλευράς του Παρατηρητηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και γι' αυτό στο όνομα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας θα πρέπει να απορρίψουμε τη συμφωνία αυτή. Σας ευχαριστώ. Κύριος Μπρόντς, παρακαλώ ένα λεπτό. Το επιχείρημα για την ε, επανεισδοχή φυσικά είναι νομικά και ηθικά αποδεκτό, αλλά γιατί πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία με το Πακιστάν για να μπορούν να πάνε στη χώρα αυτή. Θα έπρεπε να εκπλαγώ βέβαια όταν ζητάμε την ε, σύμφωνη γνώμη του Πακιστάν. Βέβαια μας λένε ότι το Πακιστάν ε, δεν συμφωνεί πάντα, ε, δεν σέβεται πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια ότι αυτό ισχύει και για τις περισσότερες χώρες του τρίτου κόσμου και για κάποιες ευρωπαϊκές χώρες επίσης. Δηλαδή όσοι είναι παράνομοι μετανάστες από χώρες οι οποίες δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να παραμείνουν στις χώρες αυτές. Αν το παραδεχθούμε αυτό γιατί να μην προσκαλέσουμε το σύνολο του πληθυσμού του Πακιστάν, της Κίνας, του Αφγανιστάν, της Μέσης Ανατολής, της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής να έρθουν όλοι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η λογική παράλογη συνέπεια αυτής της αντίληψης. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Στράσερ, 1,5 λεπτό παρακαλώ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 der Rückführungsentscheidungen auch Είμαι ευγνώμων για την ε, αξιολόγηση που θα κάνετε κυρία Μάμστον, διότι οι πραγματικές επανεισδοχές ως αριθμός είναι πολύ μικρότερος ε, από τις αποφάσεις ε, επιστροφής. 609 ήταν οι παράνομοι μετανάστες που είχαν αποφασιστεί να απελαθούν και βλέπουμε ότι έχουμε περιορισμένο αριθμό όσων επιστρέφουν. Χρειαζόμαστε μια κοινή στρατηγική στρατηγική της Ευρώπης και κοινή στρατηγική με τις τρίτες χώρες για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια Μπορσελίνο, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, η σημερινή συζήτηση για τη Συμφωνία Επανεισδοχής δεν μπορούν να αποφύγουν το ακαθόδε ζήτημα για την συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λιβύης. Γνωρίζουμε ότι ένα τμήμα της συμφωνίας επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Μας ανησυχεί το γεγονός ότι μέχρι τώρα λίγα πράγματα είπε σχετικά η Επιτροπή, παρότι η συνθήκη της Λισαβόνας επιβάλλει στην Επιτροπή να ενημερώνει ταχύτερα το Κοινοβούλιο. Όπως είναι γνωστό, η Λιβύη δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Γενέφης, ούτε μέχρι τώρα επέδειξε ότι αναλαμβάνει ε, στάση που ευθυγραμμίζεται με το διεθνές δίκαιο αφορά, τούτο αφορά και τους, ε, τους πρόσφυγες της, από την Ερυθρέα ή το κλείσιμο του γραφείου της ΥΠΑ της του ΟΗΕ. Επίσης ε, σκέφτομαι τι έγινε την περασμένη εβδομάδα όταν ένα σκάφος της Λιβύης άνοιξε πύρκατα Ιταλικού σκάφους που ήταν σε διεθνή ύδατα με την αιτιολογία ότι επάνω βρισκόντουσαν παράνομοι ε, μετανάστες. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ε, επικίνδυνη δικαιολογία που λέει ότι η συμφωνία μεταξύ Λιβύης και Ιταλίας επιτρέπει την αποπομπή την αποστολή μεταναστών στην Ιταλία χωρί το δικαίωμα να υποβάλουν έτοιμα ασύλου και την ατομική εξέταση των περιπτώσεων και που περιλαμβάνει ταυτόχρονα τη δυνατότητα χρησιμοποίηση όπλων για, την, για το σταμάτημα των, των μεταναστών. Τμήμα της συμφωνίας αυτής είναι ε, κρυφό, ξέρει το περιεχόμενο επιτροπή. Είναι αναγκαίο να ζητήσει εξηγήσει σχετικά για σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα των λιβικών αρχών να, να ανοίξουν πύρσες, σκάφη όταν υπάρχει υποψία να ε, βρίσκονται εκεί παράνομοι μετανάστες. Διότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, διακόπτει η πρόεδρος. Τον λόγο τώρα έχει... Η, ε, η κυρία Δίας Δεμέρα, ο κύριος Δίας Δεμέρα για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το άσυλο είναι μια σαφής νομική έννοια με οριοθέτηση που δεν έχει να κάνει τίποτα με συμφωνία πανεισδοχής. Η συμφωνία με το Πακιστάν είναι κοινοτικό εργαλείο που ενσωματώνεται στη μάχη της ε, καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης και όχι στο πλαίσιο της, προ... της διεθνούς προστασίας ή της παροχής ασύλου. Το αντικείμενο της συμφωνίας είναι ξεκάθαρο. Την επιστροφή Πακιστανών πολιτών που δεν πληρούν ή έπαψαν να πληρούν τις προϋποθέσεις για την είσοδο παρουσία ή παραμονή στο εδαφο ενο κρατου μέλους ή των πολιτών εκείνων τρίτων χωρών ή απάτριδων που έχουν θεώρηση ή άδεια παραμονη που έχει εκδοθεί από αρχή του Πακιστάν και εισήλθαν στο κράτος, σε ένα κράτο μέλο, νόμιμα ε, προερχόμενοι από το Πακιστάν. Σε ό,τι αφορά τον, ε, ο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου κατά τη διάρκεια του παπατισμού, πρέπει να εξασφαλιστεί μέσω τη απέτηση στήριξη των κανόνων του διεθνού δικαίου, ιδίω δε την αρχή της μη επαναπροώθησης και τον σεβασμό της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οι συμφωνίες θα εφαρμόζονται στην πραγματικότητα μόνο σε άτομα που βρίσκονται στην Ένωση παράνομα χωρίς να επηρεάζει όσους έχουν λάβει άσυλο ή έχουν ζητήσει διεθνή προστασία. Κατά την άποψή μου, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να ανακατεύουμε παρά, ε, άσχετα ζητήματα που ε, προκύπτει από την ε, επισημοποίηση ενός διεθνούς κειμένου ένωσης για τον επανατολισμό. Διακόπτει ομιλήτρια. Τελειώστε παρακαλώ. Επόμενη ομιλήτρια η κυρία Μποσκούρτ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι πλημμύρες ε, στο Πακιστάν, ε, από ό,τι φαίνεται πως προσωρινά έχουν λήξει χιλιάδες άνθρωποι, είναι βεβαίως ε, άστεγοι. Θα τους στείλουμε και τους ανθρώπους που θα επιστρέψουν στο Πακιστάν στο ίδιο αεροπλάνο με την ανθρωπιστική βοήθεια που θα στείλουμε. Αυτή η στάση έναντι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν είναι ανεύθυνη. Δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ε, επικρατεί εκεί πέρα. Δεν έχει υπογράψει καν τη συνθήκη της Γενέβης περί των προσφύγων το Πακιστάν. Πρέπει λοιπόν ε, να απαιτήσουμε είτε μια τέτοια υπογραφή είτε υπογραφή άλλων συνδικών που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό πρέπει να είναι στις συμφωνίες που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλες χώρες και επίσης να δούμε πώς θα εφαρμοστούν αυτές οι υποσχέσεις. Τι γίνεται παραδείγματος χάρη με τη συμφωνία με την Τουρκία οι διαπραγματεύσεις από ό,τι φαίνεται έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Το οριστικό κείμενο απλά βρίσκει αντίσταση από κάποια κράτη-μέλη. Μπορεί να μας πει ο Επίτροπος πού έχουν κολλήσει οι διαπραγματεύσεις. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τελειώσει αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις και αν θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα για να μπορέσουν επιτέλους ε, Τούρκοι φοιτητές και επιχειρηματίες να ταξιδεύουν χωρίς βίζα στην Ευρώπη γιατί δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για, για ελευθερία βίζα με τρίτες χώρε και όχι με μια υποψήφια χώρα. Σας ευχαριστώ τώρα η κυρία Ζίπελ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην εισαγωγική έκθεση αναφέρεται πως θα πρέπει το Κοινοβούλιο να συμφωνήσει. Δεν ξέρω αν ήταν μεταφραστικό λάθος, εγώ δεν πρέπει τίποτα. Και ακριβώς αυτή η πρώτη συμφωνία μετά τη Λισαβόνα έχει ιδιαίτερη συμβολική αξία. Ποιο μήνυμα στέλνουμε όμως εντός της Ένωσης και εκτός. Όσοι είναι υπέρ της ε, συμφωνίας μιλάνε εδώ πέρα με βάση μια βιβλική αρχή, ε, ότι εμείς νύπτουμε τα σχήρας μας και έχουμε μια σύμβαση και δεν ξέρουμε τι άλλο κάνουμε. Αλλά τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους όταν τους στείλουμε εκεί πέρα. Εγώ θα περίμενα μεγαλύτερη ευαισθησία εδώ μέσα για το τι κάνουμε με τις πρόσφυγες και για την ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ πέρα διακυβεύεται ουσιαστικά η αξιοπιστία μας όσον αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό παρακαλώ συναδέλφους να μην υπερψηφίσουν αυτή τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ κυρία Σίπελ. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Μέλτσερ παρακαλώ. Βλέπετε εδώ πέρα πως υπάρχει μια περιοριστική πολιτική όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ξέρουμε εάν μπορεί να περιοριστεί κάτι τέτοιο. Έχουμε βέβαια το παράδειγμα της Λαμπεντούζας όπου πήγαιναν, αν θέλετε, όσοι έφταναν παρανόμως στις ακτές της ε, Ιταλίας. Βεβαίως θα πρέπει, συμφωνώ, ε, να υποστηρίξουμε την υποψηφιότητα της ε, Τουρκίας. Θα πρέπει όμως να σταματήσουν παράλογες απαιτήσει όπως αυτές του κ. Καντάφου που ζητάει 5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να καταπολεμήσει τη λαθρομετανάστευση. Ανταυτού θα πρέπει τα πολλαπλά βοηθήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η αναπτυξιακή βοήθεια να συνδεθεί με την διάθεση αυτών των κρατών να καταπολεμήσουν ουσιαστικά την ε, παράνομη μετανάστευση. Επίσης θα πρέπει όσοι είναι, ζητούν άσυλο αλλά δεν είναι πραγματικοί πρόσφυγες να μπορέσουν να αποκαλυφθούν για να προστατεύσουμε ουσιαστικά τα εξωτερικά μας σύνορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στη διαδικασία και τη Το λόγο έχει ο κύριος Παπα-Νικολάου πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 80% περίπου των παράνομων μεταναστών που εντοπίζονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης ε, εντοπίζονται στην Ελλάδα στην ελλάδα το 2009 συνελήφθησαν περίπου 126.000 παράνομοι μετανάστες από αυτούς 5.000 περίπου 4.852 για την ακρίβεια ε, κατάγονται από το Πακιστάν και 36.472 από την Τουρκία. Τα αναφέρω αυτά για να καταλήξω στο εξής. Είναι πολύ σημαντική η συμφωνία με το Πακιστάν και πράγματι κράτησε πολύ, 8 χρόνια πέρασαν το άρθρο δεκαέξι προβλέπει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιμένουμε πολλά από τη συμφωνία αυτή. θυμίζω ότι σε ισπανία μάλτα ιταλία περιορίστηκαν ε, οι αριθμοί των παρανόμων μεταναστών λόγω των συμφωνιών αυτών. ελπίζω και για τη συμφωνία με την τουρκία κυρία επίτροπε να μην χρειαστούν άλλα οχτώ χρόνια. πολλέ φορέ τώρα τελευταία μα λέτε ότι βρισκόμαστε σε τελικό στάδιο δεν έχουμε όμω κάποια ανακοίνωση. ευελπιστώ και πάλι να μην καθυστερήσει πολύ περισσότερο δεν έχουμε τέτοια περιθώρια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Mr. Παπα-Νικολάου. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπα-Νικολάου. One point of clarification that doesn't seem to be very clear here. People have a status of... Μια διευκρίνηση γιατί θα μιλάμε για κάποιου που δεν έχουν εισέλθει παρανόμω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. σω είναι τούντε για άσυλο και έχει απορριφθεί αίτησή του. σω είναι κάποιοι που ήρθαν με κάποια τουριστική θεώρηση και κάτσανε παραπάνω. Οπότε δεν πρόκειται πάντοτε για κάποιου που έχουν εγκληματική πρόθεση. Αυτό είναι σαφέστατο. Το είπε η κυρία Μάλστρομ ότι θέλετε να καλύψετε τι προσδοκίε των Ευρωπαίων πολιτών. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το οποίο προσδοκά ο κόσμο στην Ευρώπη είναι να έχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σεβασμού των ανθρώπων. Ε, γι' αυτό και νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να καλυφθεί. Τώρα δεν έχω καταλάβει πώς θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε αυτού του είδους την επαναπρόθεση. Ε, πόσο το έχετε φροντίσει αυτό, από πρακτικής απόψεως, πώς θα γίνει αυτό ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Κύριος Όμπερ Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η μεγάλη εφορία για τη δημοκρατική πρόοδο της ε, Τουρκίας με το πρόσφατο δημοψήφισμα πρέπει λίγο να τη μετριάσουμε γιατί δεν συνεργάζεται καθόλου για να σταματήσει τη ροή των προσφύγων γιατί συχνά η Τουρκία αποτελεί και χώρα διαμετακομιστική των ε, προσφύγων αυτών κάτι το οποίο βεβαίως είναι απαράδεκτο το Frontex ε, πέραν των τεχνολογικών ζητημάτων δεν σημαίνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώνει για να προστατεύει τα τουρκικά σύνορα. Δεν μπορεί να μας αρμέγει εμάς συνεχώς η Άγκυρα. Θα πρέπει λοιπόν να τηρήσει τη σχετική ε, Σύμβαση για τις πρόσφυγες η Άγκυρα και θα πρέπει να δούμε τα ελλείμματα εδώ πέρα που υπάρχουν στα θεμελιώδη δικαιώματα πιέζει αφενό η Άγκυρα για στενότερες σχέσεις με τις Βρυξέλλες, από την άλλη προωθεί του ανθρώπους αυτούς στο Ελντοράντο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν να μην τρέχει τίποτα. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να ε, ολοκληρωθούν αυτές οι συμφωνίε στο ταχύτερο. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπασέσκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα στα πλαίσια της συζήτησης να μιλήσω για μια τρίτη χώρα, την Μολδόβα το 2007 το Κοινοβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Δημοκρατία της Μολδοβίας για θέματα επανεισδοχής. Ωστόσο, η πολιτική αυτή έχει κάποια κενά. Ο αντίκτυπος της πολιτικής ε, της ε, Μολδαβίας δεν έχει αποτιμηθεί επαρκώς. Οι διαδικασίες, διαπραγματεύσεις και υλοποίηση της συμφωνίας αυτής δεν ήταν επαρκώς ε, ανοιχτές κατά τη διάρκεια της κομμουνιστικής περίοδου, της κομμουνιστικής κυβέρνησης 2001 έως 9, 600.000 άτομα εγκατέλειψαν τη χώρα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τούτο ιδίω λόγω της παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη χώρα αυτή. Κάτι που αποδεικνύεται από τους, ε, τις υψηλές, τον υψηλό αριθμό καταδικών που έχει, που έχει επιβάλει το ΕΔΑΔ στην ε, Μολδαβία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ενισχύσει την ανάπτυξη της χώρας, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη χρηματοδοτική βοήθεια στη χώρα αυτή. Ο κ. Σαραλέμ Ντεζίρ. Κύριε... Αγαπητή Επίτροπε, για πρώτη φορά με το Κοινοβούλιο πρόκειται να ζητηθεί να δώσετε το πράσινο φω για μια τέτοια συμφωνία πανεισδοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντική ευθύνη που αναλαμβάνει γιατί νομίζω το Κοινοβούλιο αυτό δεν είναι δυνατόν να ασκήσει την αρμοδιότητα έτσι ε, στα ελαφρά γιατί αφορά το ε, θέμα ασφάλεια προσώπων. Ε, το Πακιστάν είναι ε, μια χώρα που δεν έχει προσυπογράψει ούτε κυρώσει τη συνθήκη της ε, Γενέβης για τους απάτριδες και τους ε, πρόσφυγες. Επομένως δεν μιλούμε τώρα για ηθαγενείς του, του Πακιστάν και για απάτριδες αλλά επίσης και για κατοίκους άλλων χωρών οι οποίοι φεύγουν από εκεί όπου μένεται ο πόλεμος και εννοώ τους Αφγανούς. Επομένως αυτή είναι η βάση συνθήκης και θέλουμε να δούμε τι θα γίνει ε, για ένα κράτος που δεν προσφέρει καμία εγγύηση, επομένως είναι θεμητό το να ζητεί το Κοινοβούλιο να γίνει μια αξιολόγηση. Αυτό άλλωστε είναι και μια δέσμευση της ε, Κομισιόν για κάποιες αντίστοιχες συμφωνίες παλιότερες και θα πρέπει το Πακιστάν να προσπογράψει πριν γίνει η συμφωνία τη συνθήκη της Γενέβης και επίσης θα πρέπει να μπορέσει να συμμετάσχει και στην αντίστοιχη επιτροπή το Κοινοβούλιο ούτω ώστε να μπορέσει να εποπτεύσει το πώς πρόκειται να συναυθεί ίσως στο μέλλον αυτή η συνθήκη. Υπ' αυτούς όρου εμείς θα δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Επίτροπο την κυρία Μάλνστρομ. Να απαντήσετε στις που Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, εξιότιμοι βουλευτές. Ευχαρίστω να συζητήσουμε για Τουρκία, Λιβύη, Μολδαβία μέσα σας, αλλά πιέζει ο χρόνος. Οπότε θα ε, επιμείνω μόνο στο κυρίως θέμα μας και κάποια άλλη στιγμή θα συζητήσουμε και τα υπόλοιπα για το Πακιστάν. Κάποιοι από τους ε, αγορητές είπαν ότι συζητούμε πάρα πολύ καιρό αυτή την συμφωνία πανεισδοχής και όλοι συμφωνούμε ότι είναι καλύτερα να υπάρχει ευρωπαϊκή συμφωνία με το Πακιστάν αντί για διάφορες σκοτεινές ασαφείς διμερείς συμφωνίες. Και αφού μιλούμε για τέτοια συμφωνία ευρωπαϊκή, μπορούμε να την εποπτεύσουμε, να την ελέγξουμε, έχει διαφάνεια, μπορούμε να τη συζητούμε εδώ στην ε, Ολομέλεια, μπορούμε να καλύψουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και επομένω υπάρχει μεγαλύτερη ασφαλή δικαίου και θα πρέπει να σας τονίσω αυτό το οποίο ήδη είπα στις αγωγές παρατηρήσεις ότι ε, το, το, το, ε, το αυτό το, δεδομένο που έχουμε που έχουμε της Ένωσης μας οδηγεί στο ε, να έχουμε ε, κατά περίπτωση ε, εξέταση κάθε ε, αιτήματο για άσυλο και υπάρχει σχετική οδηγία που θέλουμε να την αναβαθμίσουμε και έχουμε επίσης διαπραγματεύσει οι οποίε συνεχίζονται και εκεί ξεκαθαρίζονται κάποια κριτήρια για όλα αυτά και καμία συμφωνία επανεισδοχή δεν μπορεί να απελευθερώσει κανένα κράτο μέλο από αυτή την υποχρέωση. Αυτή η δήλωση που όλοι ε, προσυπογράψαμε και την υποβάλαμε στο Κοινοβούλιο πολύ σημαντική και εμείς δεσμευτήκαμε σε σχέση με τα εξή. Όπως είπαμε θα πάμε σε μια αξιολόγηση όλων των συμφωνιών επανεισδοχής και αυτή η αξιολόγηση θα είναι η βάση για μέλουσα στρατηγική, για μέλουσα επανεισδοχή και ευχαρίστω να τα συζητήσουμε και μαζί. Όσον αφορά τώρα το θέμα... Μισό να βρω τα χαρτιά μου το πώς μπορούμε να παρακολουθήσει το τι γίνεται με αυτού του ανθρώπου. Βεβαίω και δεν μπορούμε να κάτσουμε και να δούμε τι έγινε με τον καθένα από αυτού. Ούτε τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν υποχρεούνται να αναφέρουν σχετικό στην ε, Κομισιόν. Όμω αυτό θα γίνει εν ώψη αυτή τη μέλου αξιολόγηση και να δούμε πώ μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα τα κράτη-μέλη, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, όσοι επιτόπου παλεύουν τόσο ώστε να υλοποιηθούν όλα αυτά και επομένω η αξιολόγηση είναι πολύ σημαντική γιατί έτσι θα οριστεί το πώς θα διαμορφωθεί από πολιτική επανεισδοχή, αλλά αυτό δεν μας σταματήσει από το να κάνουμε βήματα πρόοδου για αυτή την συμφωνία. Και επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό με αυτή την ε, συμφωνία να μπορούμε να διαχειριστούμε την μεταναστευτική πολιτική και υπόσχομαι να επανέλθουμε για να ξανασυζητήσουμε αυτή την αξιολόγηση. Παρακαλώ αύριο να επιψηφίσετε την πρόταση. Ο Πρόεδρος, εμείς ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Και τέλος θα λέω το λόγο ο εισηγητής, ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να μην είστε πολύ αυστηρός γιατί στην πρώτη μου παρέμβαση μίλησα μόλις ε, τέσσερα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα αντί για τον κανονικό χρόνο, οπότε ελπίζω να μου αφήσετε λίγο παραπάνω χρόνο τώρα. Είναι συγκλονιστικό λοιπόν αυτό το οποίο συμβαίνει στο Πακιστάν με τις ε, πλημμύρες αλλά και με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε στο Πακιστάν είτε οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Όλα αυτά μας γεμίζουν φόβο και έχουμε βεβαίως και κάποιες αμφιβολίες για το ότι ακόμα και σε χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει τη Σύμβαση περί προσφύγων και εκεί παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και όταν ακούω συναδέλφους που είναι κατά της, ε, των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ παραβιάζουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων Σύριες τους στις χώρες ε, δεν με ευχαριστεί αυτό ιδιαίτερα και θέλω να επαναλάβω κάτι το οποίο είχα ήδη πει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλά η συμφωνία αυτή κατά κύριο λόγο δεν αφορά ανθρώπινα δικαιώματα αλλά κατά βάση μιλάμε για το ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν να αισθάνονται μια ασφάλεια και πρέπει να έχουν αυτή την ασφάλεια. Θα ήθελα να σας διηγηθώ κάτι το οποίο γίνεται στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Άστρα και ο Αμπλερ Φαρασκάν Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δικάζονταν στην ε, Μεγάλη Βρετανία και θεώρησε ένα βρετανικό δικαστήριο πως ε, εάν απελάβνονταν να κινδύνευε η ζωή τους. Οπότε έμειναν στην Μεγάλη Βρετανία. Οπότε αν είναι να απελάβνω κάποιον, καλό είναι να μην παραβιάζονται εκεί πέρα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά βεβαίω αυτό σημαίνει πως και στις χώρες μας θα πρέπει να φροντίζουμε να μην παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Πακιστάν βεβαίως έχει ακόμα πάρα πολλά να κάνει σε αυτό το τομέα και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ε, το Πακιστάν έχει και Υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και υπέγραψε φέτος ε, και κύρωσε δύο διεθνείς ε, συμβάσεις, τη Σύμβαση για Πολιτικά Δικαιώματα και Ελευθερίες και την ε, σύμβαση του 1984 η οποία απαγορεύει τα βασανιστήρια. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε αυτό. Εάν ψηφίσετε λοιπόν αύριο όχι, αυτό σημαίνει πως ε, εμπιστεύεστε μόνο τα δικαστήρια των κρατών μελών. Θέλω λοιπόν να σας ενθαρρύνω ε, να δώσετε άλλη μια ευκαιρία στο Πακιστάν μετά από 10 χρόνια διαπραγματεύσεων καθώς ε, νομίζω πως ε, βρίσκεται σε καλό δρόμο και μάλλον θα υπογράψει και τη συνθήκη της Γενέβης. Σας ευχαριστώ. Περαιούτη η συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη